Ich äh, wünsche Ihnen einen guten Morgen, insbesondere Herrn Fleckenstein. Καλημέρα σας και καλημέρα σας κύριε Φλέκενστάιν. Να δούμε λίγο. Αντιρρήσεις δεν θα υπάρχουν για την ημερήσια διάταξη, έτσι δεν είναι. Το αριθμίσαμε λοιπόν και αυτό και πάμε στο 3. Ιράν. Παρατηρήσεις. Όχι. Ψηφοφορίες. Πρώτη συμβαστική υπέρ. δώστε τον κατάλογο των ψηφοφοριών του ΕΛΚ στον Φλέκενστάιν. Κυρίε So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, συμβαστική πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 παρακαλώ υπέρ κατά απερίφθη 42 υπέρ κατά και εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 Πούντι, άνατη. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 127-128 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. ist 53 53 53-53 απερίφθη. Α, όχι, η ώρα ήταν αυτό. Καλά. 31, το σύνολο μάλλον των αριθμών 31-20. Εγκρίνεται. Λέει ο πρόεδρος. Όχι. Όχι. Καλά, αυτά καλύφθηκαν. Συμβαστική 7. Προφορικές τροπολογίες υπάρχουν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163. δύο τμήματα. Το πρώτο καταπίπτει και ψηφίζουμε το δεύτερο μόνο υπέρ. Κατά. Από και σε Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184. Ονομαστικά, λέει, γίνεται. Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό ποτέ. Preda, what I see in my EPP voting list. Να, κακό είναι να, να δούμε τον κατάλογο των α, ψηφοφοριών του ΕΛΚ. Είναι δυνατόν να έχει λάθος. Λάθος ποτέ, πάντα σωστό. Ω, ε, όχι, δεν πάει έτσι όμως, λέει ο πρόεδρος. Σκατά. The vote is opened. No, it's already long time opened back and vote. So, the vote is closed. Εγκρίνεται 34 υπέρ 20 κατά. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 186 υπέρ. Ονομαστικά και πάλι. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 24 υπέρ, 30 κατά απεριφθεί. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνατα. 197 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Παρακαλώ να σηκώνετε και τα χέρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 207 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 όχι αυτή έχει καλυφθεί 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 15 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...269. Πηδάμε δύο σελίδες. Τάνοκ. 269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Εσείς, αλλά η ομάδα έχει άλλη θέση. da. It's voting list. Look to the voting list. The vote is closed. Πέρα στις ψηφοφορίες. μία ψηφί υπέρ 35 κατά απερίφθη. 276 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 κατά αποχές εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 310 Πρώτο τμήμα το έχει καλυφθεί από τη συμβαστική 19. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Είναι σαφές εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 337. Πούντι. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 338 ε, την έχουν αποσύρει. 343. 344, συγγνώμη. Απερίφθη. Και πάμε στη συμβαστική 21, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 362, υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 439 υπέρ κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε ήταν εσείς 439 ηλεκτρονικά Ένας. 18 υπέρ, 37 κατά, 3 αποχές ε, πάμε στην επόμενη, 379 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. 381 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 389 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. 393, 393 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 405 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Και πάμε στην 22, έτσι δεν είναι. Όχι. 396 πρώτα. 396 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Και τώρα είναι η συμβαστική 22 ή ξεχάσαμε κάτι ακόμη. 395. Α, ναι. 395 γιατί απερίφθη άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 397 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 398 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 411 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 409 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 399 τώρα υπέρ κατά αποχές απερίφθη 407, 408, 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 420. Κατά, λέει ο πρόεδρος κατευθείαν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 433 τώρα παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 23 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 372 πούντι όμως λέει ο πρόεδρος. Υπέρ 372 κατά αποχές εγκρίνεται. 469 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 419 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 436-438 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 437 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 454 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 475 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 444 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 468 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 471 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ε, τροπολογία 2 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 1, υπαριθμόν 1, ε, όχι έχει καλυφθεί 3, υπέρ κατά αποχές 4, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 5 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Α, έχουμε κι άλλα Επαληθεύουμε την 24. Πέρασε. 18 υπέρ, 37 κατά, περίφθη. Και τώρα, Επιτροπή είναι η πρώτη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα υπέρ Κατά αποχές απερίφθη 5. Covered. Πάμε στην 8. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 να, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Την 11. Ελέγχουμε, επαληθεύουμε την 11. 15 υπέρ, 42 κατά, περίπου. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές. 13 δεν πρόσεχα Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συνόλο.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, δουλέψαμε πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Σας παρακαλώ όμως, μη μου φύγετε. Κύριε Φλεκερστάν, ανθρώπινα δικαιώματα είναι. Έχω τους δικούς, λέει ο κύριος Φλεκερστάν, χωρίς μικρόφωνο. So please I would like to ask you to stay here. Σας παρακαλώ να μην φύγετε.